Uh, good morning everybody. Uh, Καλημέρα σας. Ως συνήθως θα μιλήσω σου ειδικά. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο τμήμα, στο δεύτερο μέρος της ε, συνεδρίας της Επιτροπής μας. Χθες υλοποιήσαμε τις ψηφοφορίες. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο 15. Έχουμε την τιμή να μας επισκέπτεται κάποιος εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε από κοινού τις απόψεις μας για την ε, πρόσφατη εθετημένη σύμβαση. Νομίζω ότι έχει υπογραφεί από 21 χώρες. Έχει κυρωθεί μόνο από μία χώρα και αυτή είναι η Τουρκία. Δεν ξέρω πόσοι από εσά είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε το κείμενο της σύμβασης. Είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένο, μπορώ να πω. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι συμμετέχετε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή θα γνωρίζετε ότι εργαστήκαμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι η Κομισιόν ε, θα παρουσιάσει μια οδηγία για το θέμα αυτό, μάλλον για να παρουσιάσει η Κομισιόν μια οδηγία για το θέμα αυτό. Το κείμενο της σύμβασης καλύπτει πολλά από όσα θα θέλαμε εμείς να έχουμε στην νομοθετική πρόταση της Κομισιόν. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε το περιεχόμενο λοιπόν και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν σε αυτή τη σύμβαση. Και η Κομισιόν εξετάζει πώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο οργανισμός θα μπορούσε να κυρώσει τη σύμβαση αυτή. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα σας δώσω το λόγο σε λίγα λεπτά. Είχα την ευκαιρία να σας ακούσω την περασμένη εβδομάδα στην Αλβανία όπου συζητήσαμε το θέμα αυτό και πραγματικά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από το έργο σας. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να εργαστούμε εμείς ως βουλευτές για να προωθήσουμε τα θέματα αυτά και πώς μπορούν και άλλες χώρες να επικυρώσουν αυτή τη σύμβαση. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το έργο σας και θα είναι μεγάλη μου χαρά που θα σας ακούσω. Θέλω να καλωσορίσω και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και σας και τα μέλη της Επιτροπής σας που δίνετε στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, την ευκαιρία να παρευρεθεί εδώ και να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και να προωθήσουμε τα θέματα αυτά. Η ιδέα γεννήθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο όταν συζητήσαμε σε ένα γεύμα εργασίας ε, που οργανώθηκε από ένα από τους συναδέλφους στον Τιν Λάμπερτ η υποστήριξη των ε, μελών του Ευρωκοινοβουλίου εκτιμάται όχι μόνο από το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντική για να τέθει σε ισχύ συνθήκη. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σημειώσαμε τις προσπάθειές σας στον τομέα αυτό, γιατί γνωρίζουμε ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επέμεναν στο να έχουν μια σαφή αναφορά στην ε, σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και υπάρχει και μία σαφή αναφορά στο έγγραφο στην οδηγία που είναι επεκπόνηση σε σχέση με τα θύματα εγκληματικών πράξεων. Έτσι, λοιπόν, θέλουμε να συνεχίσετε να μας υποστηρίζετε στο θέμα αυτό και ξέρω ότι πρόσφατα επιστρέψατε από τα Τύρανα όπου συναντηθήκατε με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βλέπω και κάποια πρόσωπα που γνωρίζω εδώ και την κυρία Κλεβέτη, η οποία ήταν ε, αρμόδια για την προετοιμασία της σύμβασης όταν ε, μέλος της δικής μας κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Οι συνάδελφοί μας ε, θέλουν να συνεχίσουν να συνεργάζονται μαζί σας και να ανταλλάζουν πληροφορίες. Έφερα κάποια αντίγραφα του εγχειριδίου που προετοιμάστηκαν από τους δικούς μας συναδέλφους. Δυστυχώς δεν μπορούσα να κουβαλήσω πάρα πολλά αντίτυπα. Όμως είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε τρόπο να τα αποκτήσετε και Ξέρω ότι συζητάτε και με τον κύριο Μπότα για το πώς θα οργανωθούν κοινέ εκδηλώσεις για την πρόθεση της σύμβασης. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι το κοινοβουλευτικό δίκτυο της κοινέλευσης είναι ανοιχτό, μπορείτε και εσείς να συμμετάσχετε αν το επιθυμείτε. Θα μπορούσατε να γίνετε μέλη του δικτύου αυτού και να συνεισφέρετε στο έργο μας για την πρόθεση της σύμβασης είναι μία από τις προτεραιότητες για τα επόμενα δύο έτη και θέλουμε να προωθήσουμε τη σύμβαση και να διασφαλίσουμε ότι θα έχει υπογραφική κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη και πέρα από τα κράτη-μέλη και από άλλες χώρες. Δεν θέλω να σας κάνω κήρυγμα για το τι συμπεριλαμβάνεται και ποια είναι τα θετικά της σύμβασης, γιατί τα γνωρίζετε, όμως θα αναφερθώ σε κάποια θέματα που εμεί θεωρούμε σημαντικά. Καταρχήν, Πρόκειται για το μόνο νομοθετικό μέσο που υπάρχει στην Ευρώπη, νομικό μέσο που υπάρχει στην Ευρώπη για το θέμα αυτό και αφορά το θέμα της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και της ενδοικογενειακής βίας και μπορώ να σας πω ότι είναι το πιο προηγμένο σε διεθνές επίπεδο. Ε, είδαμε να εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον από άλλους διεθνείς οργανισμούς, ε, από τα Ηνωμένα Έθνη και την υπατερμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες χρησιμοποιούν τις, ε, τα πρότυπα αυτά συνεργάζονται μαζί μας για να προωθήσουν τη σύμβαση όχι μόνο στα κράτη-μέλη της Συμβουλής της Ευρώπης αλλά και στις υπόλοιπε χώρες. Η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ όταν ε, θα έχει κυρωθεί από 10 χώρες. Ε, εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να συμβεί αυτό τώρα γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ να έχουμε αυτό το πολύ καλό νομικό κείμενο, αλλά θα, παραμένει, θα παραμείνει απλώς στα χαρτιά, αν δεν κυρωθεί και αν δεν τεθεί σε ισχύ και αν δεν εφαρμοστεί από τα κρατημέλη. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε 10 κυρώσεις και 8 από αυτές πρέπει να είναι από μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η σύμβαση βασίζεται στην ε, πρόληψη, στην προστασία των θυμάτων, στη δίωξη των δραστών ε, και έχουμε και τις ολοκληρωμένες πολιτικές, ε, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ε, συμβάλλουν στην προστασία των θυμάτων. Καλύπτει τις γυναίκες ε, από όπου και αν προέρχονται, ανεξάρτητα από το, ε, από το που προέρχονται, το γενετήσιο προσανατολισμό τους, τη θρησκεία τους, το φιλί τους κτλ. Επίσης θέλουμε να καλύψουμε και άλλα θύματα ενδοκογενικής βίας και τα παιδιά αλλά και τους άνδρες, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά καλύπτει επίσης και αυτούς αλλά και τους ηλικιωμένους. Υπάρχει μια άλλη σημαντική τυχή προσπαθεί Σύμβαση να αλλάξει τις συμπεριφορές και καλή ισότητα των δύο φυλών μέσω μιας σειράς ολοκληρωμένων πολιτικών. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δίνει μεγάλη σημασία στο ρόλο των ε, εθνικών ε, οργανισμών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, τα κράτη, όταν γίνουν μέρη, υποχρεούνται να δίνουν μια ολιστική προσέγγιση στη βία κατά των γυναικών, μπλέκοντας όλους τους ενδιαφερομένους και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, τις ΜΚΟ, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δημιουργεί κάποιες, κάποια νέα αδικήματα όπως είναι η φυσική ε, και η σωματική βία, ο βιασμός, ε, έχουμε και άλλα και με όπως είναι η στήρωση, ε, ο καταναγκαστικός γάμος, εξαναγκαστικός γάμος, βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση κτλ κάποια κράτη θα πρέπει να αλλάξουν την εσωτερική τους νομοθεσία για να στήσουν νόμους για αυτά τα ποινικά δικήματα. Επίσης, ε, θα επιτρέψει τη δυνατότητα να λαμβάνονται πληροφορίες από τα κοινοβούλια, την κοινωνία των πολιτών και ε, τα εθνικά όργανα, της εθνικούς φορείς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, Έχουμε κάποια άρθρα, το άρθρο 7 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, το οποίο καλεί για πλήρεις και συντονισμένες πολιτικές και ζητά να συμπεριληφθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως ε, και τα κοινοβούλια και βουλευτές. Άρθρο 17, ε, τα εθνικά κοινοβούλια καλούνται να συμμετέχουν στην παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων ε, σε ό,τι αφορά τη σύμβαση αυτή και τα μέρη της σύμβασης θα πρέπει να υποβάλουν ε, εκθέσεις στα εθνικά τους κοινοβούλια. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε ένα σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν τα κοινοβούλια. Επίσης η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης θα καλείται συχνά να αποτιμά την εφαρμογή τη σύμβαση. Όπω σα είπα, η σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη προσπαθεί επίση να αλλάξει τι τάσει, τι συμπεριφορέ. Καλή για να υπάρξουν αλλαγέ στην οτροπία και στι εθνικέ νομοθεσίε και φυσικά τα κοινοβούλια και οι βουλευτέ θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο εκεί. Θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή νομοθεσία, να υιοθετήσουν την κατάλληλη νομοθεσία σε ε, επίπεδο ευρωπαϊκό και να είναι σίγουροι ότι γίνεται σεβαστή διεθνή νομοθεσία. Τώρα τι μπορεί να ενδιαφέρει εδώ τα κράτη-μέλη. Σήμερα 14 κράτη-μέλη έχουν υπογράψει τη σύμβαση. Αυστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Πολωνία ανακοίνωσε την πρόθεσή τη να υπογράψει πριν από τα τέλη του μήνα. Έτσι λοιπόν ελπίζουμε να φτάσουμε στον αριθμό στο 15 των κρατών μελών που θα έχουν υπογράψει τη σύμβαση. Θα πρέπει να παροτρύνεται τα κράτη-μέλη να υπογράψουν ε, και να κυρώσουν τη σύμβαση για να μπορεί να τεθεί σε ισχύ και ελπίζουμε στην υποστήριξή σας για να φτάσουμε στο μαγικό αριθμό 10. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, θεσμός πώς επεσέρχεται στην όλη εικόνα. Είμαι σύμφωνα συνάδελφος από την Κομισιόν, η Φεντερίκα θα έχει και περαιτέρω πληροφορίες. Όμως η σύμβαση είναι ανοιχτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζεται εκεί ε, στο άρθρο 75 και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την Κομισιόν ε, συνεχίζεται η εξέταση ε, το αν υπάρχει προσθεμένη αξία υπογραφής της Σύμβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συχνά ακούμε κάποια επιχειρήματα ότι τα περισσότερα από τα ζητήματα που διέπονται και ρυθμίζονται από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών περισσότερο παρά τη Κομισιόν. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτή η εξέταση και μελέτη θα μας δώσει κάποια οριστική απάντηση στο σχετικό ερώτημα. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράψει και κυρώσει τη σύμβαση, θα γίνει μέρος στη σύμβαση και επιπρόσθετα με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη θα είναι μέρη τη σύμβαση και το ίδιο θα συμβεί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν την υπογράψει και την κυρώσει. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπογράψουν και να κυρώσουν παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω μέρο τη Σύμβαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να διασφαλίσει ότι όλε οι πολιτικέ και τα προγράμματα σε πολιτικό επίπεδο συνάδουν με τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη και με τα όρια των ευθυνών τη. Εμεί τώρα υποθέτουμε ότι μπορεί να υπογράψει και να κυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε θα είχαμε ευρύτερη εναρμόνιση των μέτρων και των πρακτικών στον τομέα τη καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών και τη ενδοκογενειακή βία. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια πάτε ερωτήματα. Δεν θέλω λοιπόν να δώσω εγώ περισσότερες πληροφορίες, απλά θέλω να σας παρουσιάσω κάποια γενικά στοιχεία για το που βρισκόμαστε, για την υπογραφή και κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υλοποιείται και με εκστρατεία την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε Έχουμε την εμπειρία με τη δική μας εκστρατεία από το 2006 στο 2008 διήρκεσε και αποτελέσε τη βάση ε, για να ξεκινήσουμε την ε, κατάρτιση αυτής της σύμβασης. Σε πιο πρακτικό επίπεδο. Θα αναφέρω Κάποιες από τις εκδηλώσεις ε, που οργανώνουμε για την πρόθεση της σύμβασης μας διέπουν τρεις αρχές. Καταρχήν, να παρουσιάσουμε τις διατάξεις της ευαίσθησης, δηλαδή τι απαιτείται να κάνει το κράτη-μέλη αφού θα έχουν κυρώσει. Δεύτερο, να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σύμβαση και να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα υπογράψουν και θα κυρώσουν. Και τρίτον, να προωθήσουμε τη σύμβαση πέρα από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να υπογράψουν και να κυρώσουν, αλλά το σημαντικό είναι να το έχουν κατά νου ή να έχουν αυτή τη σύμβαση ως σημείο αναφορά όταν καταρτίζουν τη δική τους νομοθεσία ή εκπονούν προγράμματα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Επικεντρωθήκαμε σε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της σύμβασης δηλαδή είναι νομικά δεσμευτική. Όταν ένα κράτος μέλος γίνεται μέρος, δεν είναι πλέον θέμα βούλησης ε, να κάνει κάτι σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά υποχρεούται και τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν τη βία και να προστατέψουν τα θύματα και να ασκήσουν δίωξη κατά των δραστών. Το έργο της πρόθεσης μας βασίστηκε σε περιφερειακές ε, διασκέψεις. Ε, οργανώσαμε μία περσή στο Σεράγεβο όπου συναντήθηκαν οι χώρες ε, των Βαλκανίων, μία στην Πρατισλάβα, όπου είχαμε όλα τα νέα μόλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Νορβηγία, Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Και Κατόπιν πρόκειται να οργανώσουμε άλλη μία διάσκεψη στα μέσα Ιανουαρίου του χρόνου στη Φιλανδία, όπου θα συμμετάσχουν ε, όλες οι σκανδιναβικές χώρες, χώρες της Βαλτικής και Γερμανία, Πολωνία και Ρωσία. Και ξέχασα να αναφέρω ότι ήδη υλοποίησαμε μία στη διάσκεψη στη Γεωργία, στο Τίμπληση, όπου εκεί είχαμε τις ε, χώρες της Κεντρικής Ασίας και του Νοτιού Καυκάσου συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας για να διασφαλίσουμε ότι η σύμβαση θα υπογραφεί και από τα μη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν ε, ολοκληρώνεται σχεδόν ε, το έργο αυτό πρόθεση της σύμβασης και όταν θα ολοκληρωθεί θα περάσουμε σε πιο συγκεκριμένες δράσεις, δηλαδή θα προσφέρουμε αρρωγή στα κράτη-μέλη που το επιθυμούν προκειμένου να κυρώσουν τη σύμβαση και να την εφαρμόσουν. Αυτό ήταν το δικό μας έργο ως προς την προώθηση και οι δραστηριότητες αρρωγής θα λάβουν χώρα σε μεταπιτά στάδιο. Έχουμε τώρα μία κύρωση μέχρι σήμερα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν προχωρούν τα πράγματα. Σημαίνονται πρόοδο σε αρκετά κράτη-μέλη που εργάζονται προ την κύρωση. Αλβανία, Αυστρία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σερβία, Ισπανία, Σουηδία, Σλοβακία και Ουκρανία. Θα έχουμε λοιπόν μια ορμή, μια όθηση που θα δοθεί το 2013 όταν αυτές οι χώρες όταν θα έχουν ολοκληρώσει την ανάλυση της νομοθεσίας τους στο εσωτερικό επίπεδο και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις θα προχωρήσουν στην κύρωση. Μέχρι τα τέλη λοιπόν του 2013 ελπίζουμε να έχουμε σημαντικό αριθμό κυρώσεων. Χρειάζεται χρόνο για μια χώρα, είναι φυσικό μεταξύ τη διαδικασία υπογραφή και κύρωση. Ε, πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα γιατί οι χώρε πρέπει να κάνουν συγκεκριμένε αξιολογήσεις της ε, νομική του κατάστασης και των ε, οικονομικών επιπτώσεων που επιφέρει η κύρωση τη σύμβασης. Υπάρχει προφανώς κόστος και κάποιος θα πρέπει να είναι σόφρο να μην χρησιμοποιήσει την ε, πρόφαση της οικονομικής κρίσης για να μην υπογράψει ή να κυρώσει τη σύμβαση. Δεν ε, χρειάζεται να σας ε, το επισημάνω, το γνωρίζω. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές μελέτες ότι αν δεν γίνει τίποτα είναι πολύ ψηλότερο το κόστος. Θα σταματήσω εδώ και θα προτιμούσα να ακούσω τις ερωτήσεις σας αν υπάρχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν ε, ερωτήσεις ε, για πολλά θέματα. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία εδώ. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε το λόγο στους ε, συναδέλφους. Η κυρία Κλαβέτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να χαιρετήσω την παλιά συνάδελφο ε, θέλω να πω ότι σήμερα αισθάνομαι ότι είμαι σε μια ιδιαίτερα προνομιούχα θέση, καθώς ήμουν μέλος της ομάδας ε, που είχε δώσει μάχες για να πάρει σαν και ωστά αυτή η σύμβαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ήταν μια μακρά και σκληρή μάχη που τελικά είχε ένα αίσιο πέρας. Ήταν μια τεράστια μάχη που έδωσε η Επιτροπή ε, Ισότητας για το στόχο αυτό. Αυτές ήταν οι απαρχές προσπάθειες, οπότε η παρουσία σας σήμερα πραγματικά είναι ε, πολύ μεγάλη χαρά για μας. Πρόεδρε, θα συμφωνείτε μαζί μου αν πω ότι η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Γυναικών, ε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτό το θέμα. Έχουμε δώσει μάχες που να συνεχίσουμε να δίνουμε μάχες για αυτό το ζήτημα και έχουμε να κάνουμε εδώ με μία σύμβαση πολύ ισχυρή που προέρχεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μια ισχυρή σύμβαση που προβλέπει και καλύπτει θέματα όχι μόνο πρόληψης, αλλά και θέματα κυρώσεων και αντιμετώπισης και Τιμωρία τέτοιων πράξεων. Είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό το θέμα να λαμβάνουμε συγκεκριμένε και ε, ξεκάθαρες αποφάσεις, όπως παίρνουμε σε άλλους τομείς πολιτικής. Θα ήθελα να αναφερθώ πιο πολύ σε θέματα αποτελεσματικής εφαρμογής αυτής της σύμβασης μετά την υπογραφή και την κύρωσή της. Ε, γιατί σε λίγο καιρό, εντάξει υπάρχουν κάποιε καθυστερήσει, σίγουρα θα κυρωθεί και θα ε, εφαρμοστεί η σύμβαση. Οπότε τίθεται κάποια πρακτικά ζητήματα. Τα δικαιώματα των ε, θυμάτων. Ε, εγώ ε, ως δικηγόρος ε, έχω χρόνια εμπειρία στην μάχη για την προστασία των θυμάτων και για την υποχρεωτική νομική προστασία των θυμάτων. Πολλά θύματα ενδοικογενειακής βίας, κυρίως ε, γυναίκες, διότι αυτή η σύμβαση στοχεύει κυρίως τις γυναίκες θύματα, Πολλά λοιπόν θύματα δεν γνωρίζουν την νομοθεσία, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και δεν γνωρίζουν και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για αυτό το ζήτημα. Και όταν φτάνουν στο ρόλο του θύματος, δεν γνωρίζουν καν, σε κάποιες περιπτώσεις, ότι είναι θύματα και όταν συνειδητοποιούν ότι είναι θύματα δεν ξέρουν πώς αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Χρειάζεται λοιπόν μια νομική αρρωγή πρώτα απ' όλα, πέρα από άλλες κατηγορίες αρρωγής που αναφέρατε και εσείς. Κατά τη γνώμη μου η νομική αρρωγή είναι κρίσιμη σημασία εν προκειμένου. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει εγρήγορση, ενημέρωση σε όλα τα κράτη-μέλη, να υπάρχουν κατάλληλα κονδύλια για να μπορέσει να γίνει εξτρατή ενημέρωση σχετικά. Δεύτερο και σημαντικό είναι τα καταφύγια, τα κέντρα στα οποία μπορούν να καταφύγουν για βοήθεια τα θύματα. Είναι πολύ σημαντικό τα θύματα να μπορούν να βγουν από το περιβάλλον που φέρνει τη βία, όπως είναι η οικογένεια συνήθως, και να βρίσκουν κάποιο χώρο να καταφύγουν στη χώρα μου. Υπάρχουν κάποια τέτοια κέντρα, δύο-τρία ε, κέντρα, που λαμβάνουν και δημόσια χρηματοδότηση και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Όμως η χρηματοδότηση δεν αρκεί. Χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση, χρειάζονται κάποια κονδύλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα αυτά τα κέντρα υποδοχής. Το τρίτο θέμα που θέλω να αναφέρω αφορά την πρόληψη. Από τη μία υπάρχει η ελευθερία της έκφρασης. Από την άλλη υπάρχει το θέμα της ασφάλειας του ανθρώπου. Κάποιες φορές αυτές οι αρχές, αυτά τα δικαιώματα έρχονται σε σύγκρουση. Και σκέφτομαι συγκεκριμένα ένα πρόβλημα. Η πορνογραφία. Η πορνογραφία δεν είναι ποινικό αδίκημα είναι μια δραστηριότητα ένδειξη τη λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην είναι αντικείμενος πορνογραφίας ανήλικη, ώστε να μην γίνουν θύματα. Σε γενικές γραμμές όμως αυτή η δραστηριότητα θεωρείται μία ψυχαγωγική δραστηριότητα που απευθύνεται σε ενήλικες. Αν όμως δεν υπάρχουν όρια, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα με πολύ σημαντικές συνέπειες. Αναφέρουμε τώρα στο κεφάλαιο πρόληψη στο δικό σας κείμενο και αναφέρομαι στο ρόλο των ε, γυναικών στην κοινωνία εν προκειμένου. Σε τη δραστηριότητα, όπω η πορνογραφία, οι ρόλη, η κοινωνικοί ρόλοι ανδρών και γυναικών, κατανέμονται άνισα. Η πορνογραφία συνήθως χρησιμοποιεί τη γυναίκα ως κατώτερο Πιστεύω λοιπόν είναι ένα θέμα που χρήζει προσοχής και ανάλυσης. Πρέπει να ξεπεράσουμε, αν θέλετε, κάποια τέτοια όρια ε, στην, στο πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα στην κοινωνία. Αυτή η εικόνα της γυναίκας ως κατώτερο όν σε σχέση με τον άντρα είναι μια κοινωνική εικόνα που πρέπει να ξεπεραστεί και αυτό συνδέεται και με την ενδοκογενειακή βία τέλος να πω ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα ε, σε ό,τι αφορά τους μετανάστες. Διότι έχουμε μετανάστες που φτάνουν για να ζήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και έχουν ένα παρελθόν, μια κουλτούρα, μια νοοτροπία διαφορετική από τη δική μας και ε, Κάποιες φορές υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο ενδοικογενειακής βίας στον τρόπο που ζουν. Χαίρομαι γιατί διευρύνατε το πεδίο εφαρμογή ε, της έννοιας ε, της βίας και συμπεριλάβατε και τη σεξουαλική παρενόχληση ε, και άλλες ε, κατηγορίες ε, συμπεριφορών Βεβαίω, σημαίνει και το γεγονό να ασκείται βία γυναικών ακριβώ γιατί υπάρχουν κάποιε παραδόσει που τηρούν κάποιε αθλητικές ομάδε. Αυτό βεβαίω έχει τεράστιε συνέπειε. Ε, εύχομαι η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσυπογράψει αυτή τη σύμβαση και η Επιτροπή μας να δώσει μάχη για αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας και την παρουσίασή σας. Και θέλω να πω ότι θέλω να εκφράσω κάθε βούληση και διάθεση να συνεργαστώ μαζί σας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους όρους αυτής της σύμβασης. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ. Ε, συνεχίζω και σκέφτομαι γιατί υπάρχει τόση αντίσταση των κρατών μελών ε, για αυτή την ε, σύμβαση και γιατί προσπαθούν να καθησυχάσουν ε, τον κόσμο λέγοντας ότι τα κράτη προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη βία κατά των γυναικών και το συμπέρασμά μου είναι το εξής τώρα θα υπάρχει ε, όντως ένα νομικό μέσο, δηλαδή ένα μέσο προσαρμοσμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα που θα μπορεί κανείς να ε, αξιολογήσει σοβαρά και θα επιτρέψει να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών και αυτό θα αλλάξει την ισχύουσα κατάσταση γιατί βλέπουμε ότι η βία ε, στο σπίτι, στην οικογένεια δεν ε, καταλήγει απλώς στο να σκοτώνεται μία γυναίκα την εβδομάδα λόγω κακοποίησεως ε, η οποία δεν σταματά παρά μόνο όταν η γυναίκα πεθάνει και αυτό είναι φοβερό και όλοι λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει αλλά η σεξουαλική βία, η βία στην οικογένεια και η βία εναντίον των γυναικών αποβλέπουν στην ε, διατήρηση της ισχύουσας κατάστασης, της ισορροπίας των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, οι γυναίκες πατάσσονται μέσω της βίας και η κοινωνία επιτρέπει να χρησιμοποιείται η βία κατά των γυναικών οι οποίες δεν υποτάσσονται και που δεν είναι έτοιμες να δεχθούν τις ε, οδηγίες ε, και τις ε, εντολές Παραδείγματο χάρη ε, σαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είπε ότι οι γυναίκες ε, ε, θα έπρεπε να γεννούν 4-5 παιδιά αντί για ένα έως δύο και οι γυναίκες πρέπει να υποτάσσονται τότε θα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι η βία χρησιμοποιείται για να πειθαρχήσουν οι γυναίκες να υποταχθούν οι γυναίκες και αυτό είναι ο στόχος της βίας. Ε, επειδή ε, είμαι δικηγόρος, έχω ψάξει το θέμα όπως και η προλαλήσασα. Είδα λοιπόν τους φακέλους των δικαστηρίων πολλών γυναικών οι οποίες υπέκυψαν στη βία και ε, συζήτησα με θύματα βίας που επιβίωσαν και στην αρχή εξεπλάγιν. διότι υποτίθεται ότι οι γυναίκες έκαναν τόσα πράγματα στραβά, ε, ε, ήταν, ε, δεν φρόντιζαν το σπίτι τους, δεν φρόντιζαν τα παιδιά τους, δεν παρακολουθούσαν τα μαθήματα των παιδιών και την πρόοδό τους στο σχολείο ε, δηλαδή ε, υπήρχαν ε, λόγοι στην οικογένεια για τους οποίους ο άνδρας υποχρέωνε τη γυναίκα να πειθαρχήσει μέσω της βίας. Εάν λοιπόν μία γυναίκα δεν μπορεί να αναλάβει 100% την ευθύνη για όλα τα οποία συμβαίνουν στην οικογένεια, τον οικοκυριό, τον γάμο, τα παιδιά και αν δεν ακολουθεί 100% ό,τι τη ζητάει ο άντρας ή ο σύντροφό της, αν μιλάει πολύ, αν μιλάει λίγο, γιατί θα ήθελε ο άντρας αυτή να μιλάει πιο πολύ, ε, αν δεν ξέρει ακριβώς πότε ο άντρας χρειάζεται μια ζεστή σούπα, τότε ο άντρας έχει δικαίωμα να θυμώσει και να την τιμωρήσει. Εάν λοιπόν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση πρέπει να αλλάξουμε ε, την ε, ισχύουσα κατάσταση των σχέσεων ισχύω και αυτό είναι επικίνδυνο, ίσως τα κράτη το αντιλαμβάνονται και γι' αυτό ακολουθούν αυτή την οδό. Θα πρέπει όλοι λοιπόν να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη και μπορεί κάποιος από εσά να έρθει στην Ουγγαρία να μιλήσει με τους ε, βουλευτές και να τους ζητήσει να υπογράψουν διότι ούτε έχουμε υπογράψει ούτε έχουμε κυρώσει αυτή τη σύμβαση εάν όντως εννοούν αυτά που λένε για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και δεν είναι κάτι που λέγεται απλούστατα για τα μάτια του κόσμου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω απλώς ότι ζούμε σε μία πατριαρχία μια πατριαρχική δομή οικογένειας, η κυρία Βαρβάνοβα σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ε, η ιστορία που παρουσίασε η κυρία Μορβάη μου υπενθύμησε την κατάσταση της χώρας μου, της Βουλγαρίας, ε, όταν ε, εξεργαζόμουν τον φάκελο των θυμάτων εγκλημάτων που λέγεται ότι το αντρόγινο τσακώθηκε και στο τέλος ο άντρα άντρα σκότωσε τη γυναίκα του. Και τότε ο δικαστής ρώτησε τον άντρα ε, ε στη τη γυναίκα σου και τρεις φορές απάντησε ο κατηγορούμενος ναι αλλά ήταν η γυναίκα μου και ε, τελικά θώθηκε διότι σύμφωνα με το πολιτιστικό του υπόβαθρο δεν ε, ήταν κάτι που δεν μπορούσε να κάνει. Ήταν ε, μία πράξη αυτοάμυνας. Αυτή ήταν η απόφαση του δικαστηρίου. Και γι' αυτό δεν διώχτηκε σαν δολοφόνος ενός άλλου άνθρωπου. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω σχετικά με την ε, σύμβαση ότι όταν ε, καταρτίζαμε την οδηγία για την προστασία των θυμάτων χρησιμοποίησαμε τον ορισμό σας και είχαμε τη στήριξη ε, πέραν του Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορέσαμε να λάβουμε υπόψη και να περιλάβουμε την αξιολόγηση του ατόμου ψυχολογικά, ε, συναισθηματικά και να τροποποιήσουμε το δικαστικό σύστημα. Επίσης η επαγγελματική κατάρτιση και η ε, εκστρατεία συνειδητοποίησης είναι πράγματα τα οποία είναι θετικά και ευτυχώς διότι μπορέσαμε εφόσον υπήρχε αυτή η οδηγία να την ε, χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω όμως ότι το θέμα μας είναι η κατανομή εξουσίας στην κοινωνία και είδαμε ότι προσφάτως απερίφθη η πρόταση της κυρίας Ρέντινγκ για την συμμετοχή των γυναικών στα Συμβούλια των Επιχειρήσεων. Ε, απερίφθηκε από το Κοινοβούλιο και και αντιλαμβάνεστε ότι τελικά αυτή η κατανομή εξουσίας καταλήγει σε βία. Πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιον καλό τρόπο συνεργασίας όχι μόνο μεταξύ Συμβουλίου της Ευρώπης και αυτής της Επιτροπής αλλά με όλο το Κοινοβούλιο και ε, να μπορέσουμε να προωθήσουμε το νομοθετικό έργο και να στηρίξουμε την παρουσίαση της βίας εναντίον των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχασα το μικρόφωνο, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο πράγματι πρέπει να επιληθεί. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να λυθεί το θέμα αναμένοντας ε, η επόμενη γενιά να είναι πιο λογική για μένα να μην προσφεύγει στη βία. Όμως θέλω να ευστήσω την προσοχή σας σε μια άλλη πτυχή που έχει να κάνει με τη ε, κατανόηση όσο λαμβάνουν αποφάσεις. Ε, κάποιοι παραδείγματος χάρη δεν κάνουν τίποτα απλά σηκώνουν τους άμμους ε, έναντι των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν υθετούνται έγγραφα στα κράτη-μέλη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τη δική μου χώρα. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη μα, όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό, δεν βιάστηκε καθόλου για να βελτιώσει τις δικές μας νομικές πράξεις ε, και είπε υπάρχουν διάφορες παράγραφοι στα νομοθετήματα που αναφέρονται στην ε, δολοφονία κάποιου ε, εξαμιλία. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε μια ξεχωριστή νομική πράξη που αναφέρεται στη βία κατά των γυναικών. Ποια είναι η διαφορά χτυπήσει κάποιος ένα κορίτσι ή ένα γόρι. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει η ίδια αντίληψη για τη βία κατά των γυναικών σε κάθε χώρα. Έτσι λοιπόν, ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε περισσότερο αυτό το θέμα και θα έπρεπε να αναφερθούμε ρητά στο ζήτημα αυτό, γιατί σε ορισμένα κράτη-μάλλη δεν θεωρούνται ότι χρειάζονται ποσοστώσει και η χώρα της κυρίας Παρβάνοβα και η δική μου χώρα είναι στη θέση αυτή. Έτσι λοιπόν, αναρωτιούνται γιατί χρειάζεται να τα κάνουμε όλα αυτά. Όμως το 75% ε, των πτυχιούχων ε, στην Εστονία είναι γυναίκες. Τώρα θα αναφερθώ σε ένα διάσημο στον συγγραφέα, ο κύριος Τούγκλας, ο οποίος ε, το 1906 και έχει περάσει πολλούς καιρό από τότε, και δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά και έγραψε τότε δεν ε, θέλει ένας άνδρας να ε, έχει μια γυναίκα να στέκεται δίπλα του προτιμά να τα ψάχνει μόνος του τα πράγματα. Μάλιστα, κύριε Τόμσον. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω την ομιλήτρια για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δυστυχώς καθυστέρησα και δεν μπόρεσα να σας ακούσω από την αρχή. Νομίζω όμως ότι τα όσα υπόθηκαν εδώ είναι πολύ σημαντικά. Επίσης και όσα υπόθηκαν από την κυρία Παρβάνοβα επειδή ε, για αυτόν τον άνδρα που θεωρούσε ότι δεν είναι ένοχος, γιατί αυτό σχετίζεται και με την νομοθεσία. Αν η νομοθεσία δεν ε, θεωρήσει ότι είναι ένοχος, στη Δανία πριν δύο χρόνια είχαμε ένα νόμο σύμφωνα με τον οποίο αν ε, σκοτώνε κάποιος τη γυναίκα του θα ήμι τιμωρούταν και αν έδερνε τη γυναίκα του δηλαδή αν μιλάμε για κάποιον γείτονα που θα το έκανε αυτό, πάλι και αυτός θα ήμι τιμωρούταν. Σήμερα δεν μπορούμε να ε, δεκτούμε να σκοτώσει κάποιος τη γυναίκα του, ακόμη και αν μπορεί να παντρευτεί πολλές φορές. Έτσι. Λοιπόν, ε, είτε σκοτώσει κάποιος τη γυναίκα του, είτε το γείτονά του, θα πρέπει να τιμωρηθεί το ίδιο. Νομίζω όμως ότι η ισπανική νομοθεσία αναπνεύσε πάρα πολλές χώρες, γιατί στην Ισπανία είπαν «Α, ήταν γυναίκα σου». Έτσι λοιπόν, επί δύο. Η ποινή θα αυξηθεί, θα διπλασιαστεί. Και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και να σας πω πώς αντιλαμβανόμαστε το δράστη. Κάποιος ε, που χτυπά τη γυναίκα του στην Δανία θεωρείται άρρωστος. Και θέλουν να τον ε, θεραπεύσουν ενώ δεν προσφέρεται αντίστοιχη θεραπεία στη γυναίκα. Και πήγα στην Ισπανία, απευθύνθηκα στι μη κυβερνητικέ οργανώσει και ρωτήσα τι πιστεύετε για τη θεραπεία. Και μου είπαν, αυτό είναι κάτι για του αρρώστου. Και οι άντρε αυτοί δεν είναι άρρωστοι. Αν ήταν άρρωστοι, θα χτυπούσαν ε, ε, τον οδηγό του λεωφορείου, θα χτυπούσαν άλλου ανθρώπου, αλλά χτυπούν μόνο τη γυναίκα του γιατί αυτό έχει να κάνει με την κυριαρχία, με το μετσισμό. Αυτό δεν είναι αρρώστια, έτσι λοιπόν δεν είμαστε υπέρ της θεραπείας. Για τους δανούς, αυτό είναι μια σύγκρουση πολιτισμού. Γιατί εμείς ε, τους θεωρούμε ότι είναι άρρωστοι, τους θεωρούμε αρρώστους ε, και η τιμωρία είναι η θεραπεία. Έτσι λοιπόν υπάρχει ε, διαφορετική οπτική στα διάφορα κράτη-μέλη. Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσα δεν έχουν υπογράψει ακόμα τη σύμβαση. Γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση στο δικό μου κοινοβούλιο. Είπαν ότι θα υπογράψουν. Ε, ποια είναι η κατάσταση. Μπορείτε να με ενημερώσετε σχετικά. Ευχαριστούμε πολύ. Η Αντιπρόεδρος, παρακαλώ, για το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ταυτόχρονα συνεδριάζουν και άλλες επιτροπές που έπρεπε να είμαι παρούσα. Οπότε προσπαθούσα, ανάλογα με τα θέματα που συζητώ και τι υποχρεώσει που έχω, να είμαι παρούσα παντού. Σε ό,τι αφορά το θέμα τη βία κατά των γυναικών, πράγματι είναι ένα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίε μα. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μόνο θέμα ισότητας ή θέμα εξουσίας, είναι κυρίως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιο πολύ λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε το βάρος στην πρόληψη και βεβαίω στην αντιμετώπιση Με αυτή την έννοια θα ήθελα να σας επισημάνω το εξής. Για παράδειγμα, οι πολιτικές συμφιλίωσης τη επαγγελματική και προσωπική ζωή, αν ήταν οι κατάλληλε πολιτικές, θα μπορούσαν να προλάβουν την βία. Γιατί οι άνδρες αυτή τη στιγμή δεν έχουν συνηθίσει να μοιράζονται ε, τις ενδικογενειακές υποχρεώσεις, όπως έλεγε και συνάδελφο, καταλήγουν να εκνευρίζονται, να εξοργίζονται, γιατί θεωρούν ότι οι γυναίκε έχουν όλε τι υποχρεώσει μέσα στο σπίτι. Η κοινωνία επίση παραδοσιακά α, δίνει στην γυναίκα όλες τις ευθύνες για την οικογένεια, υποστήριξη στην οικογένεια, εκπαίδευση και ανατροφή των παιδιών, φροντίδα ε, στους ηλικιωμένους. Γενικότερα, όλη η οργάνωση της οικογένειας, όλες οι διαστασίσεις, είναι υποχρέωση της γυναίκας. Έπειτα, οι μισθολογικές αποκλήσεις είναι κάτι που ενισχύουν τη βία, καθώς όταν δεν υπάρχει οικονομική εξαρτησία, οι γυναίκες πολύ συχνά εξαρτώνται και ε, υποτάσσονται στον άντρα. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ειδική κατάρτιση για τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές, διότι θα πρέπει να γνωρίζουν να ερμηνεύουν ήδη τα πρώτα σημάδια, τα, ε, τα πρώτα αν θέλετε, όντως ένα γερμό που θα πρέπει να χτυπήσει όταν βλέπουν, αν θέλετε, κάποια κρούσματα. Π.χ. την πρώτη καταγγελία. Μια καταγγελία που δεν αξιολογείται πολλές φορές καταλήλως και η γυναίκα τελικά παραμένει απροστάτευτη. Επιστρέφει σπίτι, η βία συνεχίζεται και τελικά μπορεί να καταλήξει στο θάνατο. Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές αρχές, θέλω να πω ότι η πορτογαλική νομοθεσία είναι πολύ καλά. Δηλαδή, το, η βία, η ενδοικογενική βία θεωρείται αυταπάγγελτα α, διώξιμο ε, αδίκημα, δηλαδή δεν χρειάζεται να υπάρξει καταγγελία. Αναλαμβάνουν α, αυταπάγγελτα οι διοκτικές αρχές. Όμως, να πω το εξής. Να σας αναφέρω μια πρόσφατη δικαστική απόφαση. Ένας δικαστής αποφάσισε ότι η ποινή για ενδοικογενειακή βία ήταν ο κατοίκον περιορισμός. Δηλαδή, να μείνει στο σπίτι αυτό ο και να συνεχίσει να χτυπάει τη γυναίκα του. Αντί δηλαδή να απαγορεύσουν στον θήτη να πλησιάζει το θύμα, όπως συνήθως συμβαίνει, αυτός ο δικαστής που φαίνεται ότι έχει μια πολύ ιδιαίτερη ε, άποψη για την κοινωνία, έδωσε ως ποινή τον κατοίκον περιορισμό. Βεβαίω η κατάσταση επιδεινώθηκε. Και σε αυτή την περίπτωση, ναι, ναι, δεν βρήκε το θάνατο η γυναίκα, αλλά ε, βρίσκεται σε πολύ δινή κατάσταση. Χρειάζεται λοιπόν κατάρτιση. Πρέπει να επενδύσουμε στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση των αρμόδιων φορέων, των διοκτικών αρχών, αστυνομία και δικαστικές αρχές. Επίσης χρειάζονται ενημερωτικές εκστρατείες στις γυναίκες για τα δικαιώματά τους. Και επίσης πού μπορούν να προστρέξουν, ε, τι δικαιώματα και δυνατότητα τους δίνει η ίδια η κοινωνία. Έπειτα, σε ό,τι αφορά και πάλι την αντιμετώπιση της κατάστασης, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα βίας, πώ τα αντιμετωπίζουμε. Πέρα από την νομοθεσία, που θα πρέπει να έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία, χρειαζόμαστε και προστασία του θύματος από όλες τις απόψεις. Οικονομική προστασία, νομική προστασία, ψυχολογική υποστήριξη, όλες λοιπόν τις μορφές υποστήριξης προς το θύμα, και όταν εμπλέκονται και ανήλικοι, παιδιά, εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες για να συνεχίσουν να ε, βιούν ε, τα παιδιά με την μητέρα. Όταν δηλαδή πολύ συχνά οι γυναίκες θα πρέπει να καταφύγουν σε ε, ένα κέντρο υποδοχής, όπως συμβαίνει και στη χώρα μου. Έχουμε διαπιστώσει ότι Πέρα ότι πολύ συχνά είναι και τα τα παιδιά θύματα της βίας και ψυχολογικά φθύρονται πάρα πολύ από τέτοιου είδους εικόνες και γεγονότα, από αυτά που βλέπουν, αλλά και όταν απομακρύνονται από τη μητέρα τους. Τέλος, να πω ότι είναι προφανές ότι ε, στη σημερινή, η σημερινή κατάσταση οικονομικής ε, κρίσης, κοινωνικής κρίσης, συνεχών πιέσεων, πιέσεων ψυχολογικών μέσα στην οικογένεια, περικοπών στις δημόσιες δαπάνες της υγείας, άρα ε, βλέπουμε ανθρώπους που πιέζονται, πιέζονται οικονομικά και πιέζονται και ψυχολογικά οι άνθρωποι. Όλα αυτά συμβάλλουν εξίσου σε ένα αρνητικό κλίμα, κάποιες φορές εκρηκτικό κλίμα μέσα στην οικογένεια. Φανταστείτε σε κατάσταση ανεργίας, άγχους, στρες, όλα αυτά ενισχύουν την εκδήλωση βίας. Πρέπει λοιπόν να δοθεί προτεραιότητα από μας, από εδώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον τομέα έχει κάνει πολύ σημαντικές μελέτες. Άρα, από κοινού θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια πληγή, διότι έχει τεράστιες άμεσες και μακροχρόνιες συνέπειες για την όλη κοινωνία μας και βεβαίως προκαλεί θύματα. Διότι ο αριθμός των θυμάτων των θανατηφόρων, ε, αν θέλετε, κρουσμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά. Μιλάμε για θανάτους. Θανάτους γυναικών από τους συντρόφους και τους συζύγους. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ζήτηση που πρέπει να συνεχίσουμε. Θα πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να κυρώσουν αυτή την σύμβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Γκαρθία Πέρες έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, όπως και η σύντροφος, γιατί και εγώ στο συγγνώμη που δεν ήμουν παρούσα από την αρχή της συνεδρίασης. Πράγματι έχουμε πολλές αρμοδιότητες και συνεδριάζουν διάφορες επιτροπές. Όμως αυτή τη στιγμή συζητούμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ήταν αντικείμενο συζήτησης και εργασίας της Επιτροπής μας και στο παρελθόν. Και ακολουθώντας την ε, προσέγγιση της ΕΔΙΤ, θέλω να πω και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε όλοι ότι το φαινόμενο της βίας κατά του φύλου είναι ένα οριζόντιο ε, πρόβλημα και θα πρέπει λοιπόν να παρέμουμε παντού. Είναι μία κοινωνική πληγή αυτή η βία. Και βεβαίως συμβαίνει σε μία άνεση κοινωνία. Γεννάται λοιπόν μέσα από την ανισότητα. Όταν ένας άνθρωπος έχει περισσότερη εξουσία και πιο πολλά δικαιώματα από τον άλλο, έτσι γεννάται η βία. Αυτό είναι ιστορικά κάτι που μπορούμε να αποδείξουμε. Αυτό επίσης που πρέπει να πούμε είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να αρχίσουν να δουλεύουν πάνω σε αυτό το θέμα. Η αντιμετώπιση της βίας ε, κατά του φύλου είναι ένα οριζόντιο ζήτημα που πλήττει μία σειρά πολιτικών. Χρειάζονται λοιπόν πολιτικές διαφορετικές, άμεσα και μακροπρόθεσμα για να αντιμετωπίσουν ολοκληρωτικά το φαινόμενο. Δυστυχώς, οι θεσμοί είναι δυσκίνητοι. Τα αποτελέσματα δεν φαίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη προσπάθεια και μακροχρόνια προσπάθεια. Χρειάζεται λοιπόν από τη μία πολιτικές προστασίες και υποστήριξη των θυμάτων, όπως έλεγε και η Μπρίτα. Η Ισπανική νομοθεσία, για παράδειγμα, προσφέρει αποφασιστική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας. Α, πρόκειται για ποινικά αδικήματα εγγεγραμμένα στον ποινικό κώδικα Αλλά από εκεί και πέρα μπαίνει και το ζήτημα της μετέπειτα επανενσωμάτωσης ε, στην κοινωνία. Δηλαδή για να μπορέσει ξανα, να επιστρέψει στην κοινωνία κανείς, στην αγορά εργασία στην, στην κανονική ε, ζωή, ε, για να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι, να μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά τους, χρειάζονται κάποια υποστήριξη και κυρίως οικονομική υποστήριξη. Χρειάζονται λοιπόν και αυτά τα μέτρα παράλληλα με την πρόληψη επειδή στην κοινωνία μας υπάρχουν πολλές ανισότητες, θα πρέπει ήδη να σκύψουμε πάνω στα παιδιά μας, τα παιδιά μας, τα αγόρια μας, τα κορίτσια μας, από τώρα να τα νουθετήσουμε τον κατάλληλο τρόπο, ώστε αργότερα, όταν θα μεγαλώσουν, να μην αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο της βίας. Χρειάζεται λοιπόν η σωστή ανατροφή. Είτε μιλάμε για εκπαίδευση στο σχολείο, καθώς και οργανώσεις που ασχολούνται με αυτό το θέμα μπορούν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μας, γιατί θα πρέπει από μικρά τα παιδιά μας να γαλουχηθούν με γνώμονα την ισότητα. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί σήμερα να μεγαλώνει πιστεύοντας ότι μεγαλώνοντας θα μπορεί να επιτεθεί στη σύντροφό του απλά και μόνο γιατί είναι άντρας. Χρειάζονται λοιπόν πολιτικές όχι πυροσβεστικέ, δηλαδή απλά να προσφέρουν υποστήριξη στη γυναίκα που είναι θύμα βία, το οποίο είναι θεμελιώδε, βεβαίω. Και ήταν σημαντική αλλαγή αυτή που έγινε τα τελευταία χρόνια και πρέπει να το αναγνωρίσουμε στη χώρα μου. Πριν από 15 χρόνια η γυναίκα δεν αποφάσισε να πάει να καταγγείλει στι αρχές μια τέτοια πράξη βίας. Γιατί πολύ συχνά και η αστυνομία τι έλεγε. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι οικογενειακά, είναι προσωπικά ζητήματα. Πάτε σπίτι σας και βρείτε τα με τον άντρα σας. Αυτά, αυτά λεγόντουσαν. Αυτά γίνονταν στο παρελθόν. Καταφέραμε, πιστεύω, να ξεριζώσουμε αυτές τις νοοτροπίες σήμερα. Δύσκολα μπορεί να δικαιολογήσει κανεί μια τέτοια πράξη βία, λέγοντα «Ε, εντάξει, και η γυναίκα αυτή εκνεύρισε τον άντρα τη. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Αυτό από τη μία πλευρά και από την άλλη τα μέτρα πρόληψης ε, και παιδείας, σωστής ανατροφής των παιδιών. Και βεβαίω πρέπει να εγκαλέσουμε τα κράτη-μέλη, να εγκαλέσουμε τις κυβερνήσεις και να εγκαλέσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει. Να προχωρήσει όχι μόνο στην νομισματική πολιτική και σε οικονομικές πολιτικές, αλλά και σε άλλες πολιτικές στις πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολιτικές ε, που δίνουν ε, σημασία στις ε, βασικές αξίες του ανθρώπου. Η αρχή συγγνώμη, της ισότητας είναι από τις βασικότερες αρχές που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέματα που έχουμε θέσει όλες μας εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχουμε καταφέρει να, τελικά να έχουμε μια οδηγία με αυτό το θέμα. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να υπάρξει μια, αν θέλετε, τυποποίηση, να υπάρξει μια κωδικοποίηση όλων αυτών των φαινομένων και να χαρακτηρίζονται όλες αυτές οι πράξεις ποινικό αδίκημα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να δεσμευτούν τα κράτη-μέλη ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να μην υπάρχει στο μέλλον. Έχουν γίνει πολλά στο παρελθόν, στα τελευταία χρόνια, αλλά πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να αγωνιζόμεθα. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο του Συμβούλου της Ευρώπης που ήρθε να κάνει αυτή τη ζήτηση μαζί μας. Και αν μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, είμαστε στη διάθεσή σας. Eh, Ευχαριστώ. Και δίνω τώρα τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πριν από αυτήν στην κυρία Κουτλάσκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη έχουν ε, λεχθεί μέχρι στιγμής. Εκπροσωπώ μία από τις χώρες οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογράψει την ε, συνθήκη έχει συζητηθεί όμως το θέμα πάρα πολύ ε, στα μέσα ενημέρωσης και ε, εκ των υστέρων η κυβέρνηση απεφάσισε να ε, προσυπογράψει αυτή τη συνθήκη και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ποιος ήταν ο λόγος αυτής της καθυστέρησης και της εναντίωσης στη συνθήκη ήταν το άρθρο 12 Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν το άρθρο αυτό, το άρθρο 12, προκαλεί τέτοιες αφισβητήσεις και σε άλλα κράτη-μέλη και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο δεν έχει ε, υπογραφεί και από άλλα κράτη αυτή η ε, συνθήκη όπως ε, ήταν η περίπτωση στην Πολωνία. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι και χαίρομαι ιδιαίτερος διότι ο λαός ε, ήταν ε, λογικός και στη συνέχεια η κυβέρνηση και ε, η Πολωνία λογικεύτηκαν και είναι έτοιμοι τώρα να υπογράψουν. Αλλά ήθελα να ρωτήσω αν το άρθρο 12 είναι τόσο αμφιλεγόμενο και κατέληξε στο να μην θέλουν να την υπογράψουν. Και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην εκπρόσωπο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο Καταρχήν, θα ήθελα να επανέλθω σε ορισμένα χαρακτηριστικά και να σας πω ότι ε, αυτή η σύμβαση είναι το πρώτο ε, δεσμευτικό μέσο που προστατεύει τις γυναίκες ε, εναντίον της βίας με αποτελεσματικά μέτρα. Επίσης ε, περιλαμβάνει και έναν ορισμό του φύλου που είναι επίσης πολύ σημαντικό καθορίζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, εξασφαλίζει ότι τα κράτη θα λάβουν, που συμμετέχουν και προσπογράφουν θα λάβουν όλα τα μέτρα για να καταπολεμήσουν αυτή τη βία, τη βία κατά των γυναικών, την ε, ε, βία στην οικογένεια εναντίον των γυναικών και των παιδιών και την βία στην κοινωνία. Ε, όπως ε, ε, είπε και το Συμβούλιο της Ευρώπης θέλουμε να ενισχύσουμε την καταπολέμηση της βίας εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, υπάρχει θέληση αυτή δεδηλωμένη μέσω διαφόρων ε, νομοθετημάτων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών που θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα εμπόδιο στην ισότητα των φύλων. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα νομικά δεσμευτικό μέσο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναιτών ιδίως εις τα πλαίσια της οικογενείας έχουμε διάφορα νομοθετήματα αλλά κανένα με την ίδια εμβέλεια με αυτή την σύμβαση. Ε, όπως ε, είπε η συνθήκη τη, ε, ε, όπως είπε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης το άρθρο 75 παράγραφος 1 προβλέπει ότι θα πρέπει να υπογραφεί όχι μόνο από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον των κρατών μελών και όχι εν ονόμα των κρατών μελών και το τονίζουμε αυτό και γιατί. Παραδείγματο χάρη, διότι υπάρχουν πολλές ποινικέ διατάξεις ή στη συνθήκη αυτή και επ' αυτόν μόνο τα κράτη έχουν, ε, είναι εξουσιοδοτημένα να δράσουν Παραδείγματο χάρη οι κατηγορίες τη της όπου η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί ε, να ε, περιγράψει τις διάφορες ε, μόρφες της βίας κατά των γυναικών, υποχρεωτική στήρωση, ακροτηριασμός των γεννητικών οργάνων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμως ε, δεν είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ε, στα θέματα αυτά έχει συμφωνήσει να υπάρχει ελάχιστη εναρμόνιση, δηλαδή εάν δούμε το κεφάλαιο που αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων βλέπουμε ότι ε, η βάση είναι το άρθρο 81 και 82 της συνθήκης. Ξέρουμε ότι η αρμοδιότητα αυτή έχει εξαστηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίως μέσω διαφόρων ε, νομικών ε, πράξεων εκ των οποίων ε, το πιο πρόσφατο είναι η οδηγία η οποία αναφέρεται στα ελάχιστα πρότυπα για τη στήριξη στα θύματα της βίας. Αυτό σημαίνει... on minimum η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν έχει άμεση αρμοδιότητα και τα κράτη-μέλη πρέπει με τη σειρά τους να καταρτήσουν μηχανισμούς για να εφαρμόσουν τη συνθήκη άρα υπάρχει συμμετοχή ε, και των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε τομείς όπου υπάρχουν ε, ορισμένες ε, αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και γι' αυτό αιτιολογείται η προσυπογραφή και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών μελών χωρίς αυτό να είναι μία υποχρέωση, είναι μία πολιτική επιλογή κατόπιν των αναλύσεων των νομικών επιπτώσεων και της προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο της Ενώσεως εξού και επιβεβαιώνω ότι η ανάλυση όλων των νομικών επιπτώσεων <clears throat> αυτή τη στιγμή εξετάζεται ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας αυτό στο τέλος του έτους. Ουσιαστικά Θέλουμε να εντοπίσουμε τις αρμοδιότητες ε, για να υπάρξει μία ευρωπαϊκή νομοθεσία να αναθυθεί λυθεί η αρμοδιότητα αυτή στα πλαίσια και από τη σκοπιά αυτής της σύμβασης, να δούμε ε, πού είναι ε, αρμόδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχει εξασκήσει ακόμη την εξουσία που διαθέτει. Βλέπουμε ότι 14 κράτη-μέλη μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει τη συνθήκη, αλλά δεν την έχουν ακόμη ε, κυρώσει. Οπότε αυτό είναι ε, ενδεικτικό ότι ε, το θέμα είναι περίπλοκο και μπορεί να είναι αμφιλεγόμενο όπως απεδείχθη κατά τη διαπραγμάτευση του κειμένου και κράτη-μέλη μεμονωμένα ε, δεν θα προσχωρήσουν ή ε, θα διατυπώσουν επιφυλάξεις σχετικά με το άσυλο και την άδεια παραμονής ε, για τους άντρες, γυναίκες και παιδιά. Δέχεται λοιπόν η σύμβαση αυτή να να μην, να μην τύχεις της προσχωρήσεως Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μία πρόταση για απόφαση στα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο και βεβαίως τα κράτη-μέλη στην περίπτωση αυτή θα μπορέσουν να επηρεάσουν τον ή όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα α, υιοθετηθεί. Βλέπουμε ότι ε, θα πρέπει να υπάρξει μία πράξη ε, για την προσχώρηση και την κύρωση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ενδεχομένω ε, ε, ένα άλλο χρήσιμο μέσο θα ήταν μία δήλωση αρμοδιότητος που θα αποτελέσει παράρτημα στην απόφαση του Συμβουλίου τονίζοντας ότι η κατανομή των εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένη και αυτό μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμο για να μπορέσει να διευκολύνει την περαιτέρω παρακολούθηση και υποβολή στοιχείων στον μηχανισμό ελέγχου της εφαρμογή συμβάσεως στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα ολοκληρώσω εδώ και είμαι στη διάθεσή σας για να σας δώσω περαιτέρω εξηγήσεις αν θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλέσαμε επίσης ε, και εκπρόσωπο από την ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο τώρα στην ε, εκπρόσωπο της ΕΟΚΕ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Ήταν πολύ διαφωτιστικά τα όσα ακούστηκαν ε, και μπορώ να σας πω ότι η δική μας Επιτροπή για πολλά χρόνια παρακολουθεί το ζήτημα της ε, ισότητας μεταξύ των δύο φύλων της ενδοκογενειακής βίας, της βίας κατά των γυναικών. Και μόλις την περασμένη εβδομάδα, μάλλον αυτή την εβδομάδα, εγκρίναμε ένα έγγραφο σχετικά με την ε, ενδοκογενειακή βία και θέλω να ευχαριστήσω εδώ τους ομιλητές γιατί θα παρευρεθούν αύριο μαζί μας γιατί έχουμε μια ειδική διάσκεψη στο κτίριό μας στην ε, Οδό Μπελιάρ για το θέμα της ενδοκογενικής βίας. Θέλω να αναφερθώ σε κάποια σημεία που εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή αυτής της πολύ σημαντικής ε, σύμβασης. Θα είμαι σύντομη. Το πρώτο που θέλω να θέσω είναι πώς ε, πώς ε, θα αναγκάσουμε την αστυνομία να λογοδοτήσει αν ε, δεν επιτελεί το καθήκον της όπως πρέπει και μπορώ να σας πω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο πολύ συχνά έχουμε το θάνατο του θύματος ε, ως αποτέλεσμα πώς λοιπόν θα λογοδοτήσουν όταν υπάρχουν καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες και μπορεί να έχουμε το θάνατο των θυμάτων Όταν ε, μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία, αυτή καλύπτει και σχέσεις ε, όταν συζούν τα άτομα ή μπορεί να μην έχουν συζήσει ποτέ τα άτομα στο ίδιο σπίτι ή δεν ζουν πια στο ίδιο σπίτι. Δηλαδή χρειαζόμαστε πάρα πολύ προσεκτική νομική διατύπωση για να καλύψουμε το θέμα αυτό διαφορετικά όπως συμβαίνει και σήμερα στην εθνική νομοθεσία, υπάρχουν πάρα πολλά κενά, πάρα πολλά παραθυράκια στην νομοθεσία και πρέπει αυτό να το επιλύσουμε. Και κάτι ακόμη, το θέμα του να έχουμε επαγγελματίες ε, που θα προσφέρουν αρρωγή στα θύματα θα βοηθούν τα θύματα να έχουν ε, πρόσβαση στη βοήθεια που χρειάζονται. Επίσης, έχουμε και το θέμα της ιδιωτικής ζωής. Ε, πώς θα τα επιλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Και θα ολοκληρώσω εδώ, απλά θέλω να κάνω το εξή σχόλιο. Πρέπει να ε, καλύψουμε και τους νέους, ακόμη και τους εφήβους σε αυτές τις καταστάσεις. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ομιλήτρια, την προσκεκλημένη μας, για να συνοψίσει κατόπιν όσων ακούστηκαν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπήρχε ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε σε όλες τις περιβάσεις ε, για την ε, έλλειψη ισότητας μεταξύ των δύο φύλων ε, και μια έκκληση για να αλλάξουν νοοτροπίες και καλύτερη παιδεία κυρίως για τα γόρια και τους άνδρες προκειμένου να αλλάξουν τα μοντέλα συμπεριφοράς. Αυτό είναι ένα, αυτή είναι μία από τις κύριες διατάξεις ε, της Σύμβασης. Ανέφερα προηγουμένως ότι πρόκειται για μία νέα έκκληση για περισσότερη ισότητα και για μία αλλαγή ε, στην ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να υπάρξουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικές εκστρατείες, όμως φυσικά πρέπει να καλούμε για περισσότερη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, γιατί εν τέλει η βία βρίσκεται ρίζες στην ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Αυτό αναφέρθηκε πάνω κάτω από όλους όσους πήραν το λόγο. Η κυρία Κλεβέτη επίσης αναφέρθηκε στο εξή ζήτημα, αν η σύμβαση καλύπτει άλλα ζητήματα όπως την προστασία των μεταναστών. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένε διατάξεις στη σύμβαση που έχουν να κάνουν ε, με την προστασία των μεταναστριών. Έτσι λοιπόν θα σας συνιστούσα να εξετάσετε την ιστοσελίδα μας. Έχουμε κάποια θεματικά έγγραφα όταν ε, μιλάμε για τη σύμβαση και τα παιδιά, τη σύμβαση και τις μετανάστριες, ε, τη σύμβαση και το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων κτλ. Θα συνεχίσουμε να εκπονούμε τέτοια θεματικά έγγραφα και να τα βάζουμε στην ιστοσελίδα μας. Θα είναι διαθέσιμα λοιπόν ηλεκτρονικά και φυσικά αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας καθώς θα συνεχίσουμε να ελοποιούμε συγκεκριμένες μελέτες που σχετίζονται είτε με συγκεκριμένα άρθρα της σύμβασης ή θεματικές μελέτες. Θα βρείτε λοιπόν αρκετές πληροφορίες ήδη. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα σχετικά με τις διατάξεις, ε, αλλά σίγουρα καλύπτονται και οι μεταναστές και τα παιδιά από τη σύμβαση. Σε ό,τι αφορά τώρα την παρέμβαση της κυρίας Μορβάη και εσείς αναφερθήκατε στη στάση, στην αλλαγή στάσης και νοοτροπίας και γιατί υπάρχει ε, ουσιαστικά από κάποια κράτη-μέλη αντίσταση σε αυτό. Όπως σας είπα, συνεχίζουμε το έργο μας σε αυτήν την κατεύθυνση. Η κυρία Περβάνοβα αναφέρε ε, το πολιτιστικό background. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ένα από τα συγκεκριμένα σημεία της σύμβασης είναι ε, έκκληση για αλλαγή νοοτροπίας ε, και κουλτούρας. Εδώ μιλάμε για κάποιες διατάξεις της σύμβασης που καλύπτουν τα εγκλήματα τιμής. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τους δράστες. Τώρα για τη δέσμη μέτρων για τα θύματα. Εξετάσαμε τα έγγραφα, τα πιο πρόσφατα έγγραφα συνάδουν αρκετά οι διατάξεις αυτές με τις διατάξεις σύμβαση δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ του πακέτου της Κομισιόν και της σύμβασης, όμως προχωρούμε λίγο παραπέρα σε ό,τι αφορά στον καλύτερο ορισμό της ενδοκογενειακής βίας και χαίρομαι που αναφέρθηκε αυτό από αρκετές ομιλήτριες γιατί συχνά έχουμε πρόβλημα στη μετάφραση στις διάφορες γλώσσες Έχουμε ένα φυλάδιο ήδη επιγραμμικά σε πάνω από 20 γλώσσες που παρουσιάζει και συχνά η ενδοκογενειακή βία ε, ουσιαστικά μεταφράζεται ως βία μέσα στην οικογένεια. Όμως ε, δεν σημαίνει μόνο αυτό, πηγαίνει παρατέρα. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν ζει κάποιος κάτω από την ίδια στέγη. Μιλάμε για στενές σχέσεις και έχουμε πρόβλημα γιατί η μετάφραση είναι λάθος στις περισσότερες γλώσσες και πρέπει να το δούμε αυτό. Ορισμένα κράτη-μέλη αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καν ορολογία. Προσπαθούν τώρα να την εξεύρουν, ξέρω ότι στην Νορβηγία μόλις ε, κατέθεσαν κάποια νομοθεσία που ουσιαστικά αναφέρεται στη βία μεταξύ ανθρώπων που έχουν στενές σχέσεις και όχι στην ενδοοικογενειακή βία. Σας ευχαριστώ όμως που το επισημάνατε αυτό και κάθε φορά που έχετε ευκαιρία να το αναφέρετε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου. Επίσης, Ακούσαμε ότι κάποιες χώρες δεν ε, έχουν ε, σκοπό να ασχοληθούν με το θέμα της σύμβασης. Ε, δεν είναι καν στην ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό. Το ακούσαμε για την Εσθονία. Ακούσα ότι ε, περιγράφουν κάποιους ανθρώπους που επιδιώκουν ε, την υλοποίηση τη σύμβαση ω ε, τρέλε φεμινίστριε. Κοιτάξτε, άκουσα και το σχόλια την Πολωνία. Πρέπει να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη. Δεν μιλάμε για μια ιδεολογία τρελών φεμινιστριών. Θέλουμε να προστατεύσουμε τι γυναίκε από τη βία. Ήταν δύσκολη η συζήτηση. Η Λιθουανία ήταν μία από τι χώρε όπου πήγαμε στο κοινοβούλιο και είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων όχι μόνο δεν είναι στην ημερησία διάταξη το θέμα αυτό και μάλιστα οι βουλευτές μας το είπαν περισσότερο και όχι τόσο η κυβέρνηση, αλλά μας είπαν ότι δεν σκοπεύουν να ασχοληθούν με το ζήτημα ούτε στο εγγύς μέλλον. Και ενώ κάποιες χώρες προχωρούν ε, και υπογράφουν και κυρώνουν τη σύμβαση, κάτι τέτοιο θα μας βοηθήσει να παρουσιάσουμε την πρόσθετη αξία, την προσθέμενη αξία της σύμβασης σε όσους αντιστέκονται περισσότερο. Η Δανία είναι μία από τις χώρες, επίσης έχουμε δυσκολίες, δεν ε, υπήρχαν ε, πολλές πληροφορίες από τη Δανία. Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ στην Ισπανία, αναφέρθηκε ως ε, ένα καλό παράδειγμα η σύμβαση. Δεν είναι μία εξωπραγματική εφεύρεση, ουσιαστικά αποτελεί μία ομαδοποίηση βελτιστών πρακτικών. Έτσι λοιπόν οι νομοθέτε τι προσπάθησαν να κάνουν, να ομαδοποιήσουν τι ε, καλέ εμπειρίε και την νομοθεσία από τα κράτη-μέλη, απλώς σε ένα υψηλότερο επίπεδο για να έχουμε αυτό το νομοθέτημα. Δεν έρχονται λοιπόν όλα αυτά από το πουθενά. Πρόκειται για ένα κείμενο που βασίζεται στι τρέχουσε πρακτικέ και υπάρχουν βελτιστέ πρακτικέ στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε ότι δεν πρόκειται για ένα κείμενο που έρχεται από το μηδέν, αλλά υπάρχουν παραδείγματα στα κράτη-μέλη και τα έχουμε βάλει από κοινού προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτές τις βαλτέ πρακτικέ. Η κυρία Στρέλα αναφέρθηκε στην ενισότητα, στη σημασία της εφαρμογή και τι θα κάνουμε με την επιβολή του νόμου. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις, ε, δεν είναι μόνο θέμα καλής για το αν τα κρατημέλη ε, θα γίνουν μέρη της σύμβασης. Δηλαδή πρέπει να βρουν ε, και τα απαραίτητα κονδύλια και για την κατάρτιση της αστυνομία, των δικαστών, των εισαγγελέων. Θα πρέπει λοιπόν να εξεύρουν κονδύλια προκειμένου να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να καταρτήσουν τους αστυνομικούς για να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις ενδοκογενικής βίας και βίας κατά των γυναικών. Γι' αυτό και πάλι το τονίζω, είναι σημαντικό να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση και στη συνέχεια τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν συγκεκριμένα μέτρα. Κυρία Καρσιά Πέρες, αναφέρεται τη σημασία των ολοκληρωμένων πολιτικών. Εγώ αναφέρθηκα ε, στο τέταρτο πυλώνα όπως ε, το ονόμασα, τις ολοκληρωμένες πολιτικές, δηλαδή πρέπει οι δικαστές οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αστυνομικοί και άλλοι μοντινά συνεργαστούν, ε, κυρίως όταν μιλάμε για την προσφορά υπηρεσιών στα θύματα και σε ό,τι αφορά την παροχή καταφυγίων και τη διαχείριση, τη δίκηση των καταφυγίων αυτών. Θα κάνω ένα σχόλιο. Πολύ ωραία να μιλάμε για την νομοθεσία, για τα προγράμματα. Αλλά τι πρέπει να έχουμε κατά νου, ότι η σύμβαση προβλέπει ένα πολύ συγκεκριμένο, πολύ ολοκληρωμένο σύνολο νομικών μέτρων και άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν πρέπει να προωθήσουμε την υπογραφή και κύρωση της σύμβασης. Χρειαζόμαστε πολιτική βούληση. Δεν είναι ότι τώρα δεν έχουμε κανένα νομοθέτημα, έχουμε ένα κείμενο ή είναι κείμενο, είναι θέμα πολιτική βούληση η υιοθέτηση και εφαρμογή αυτού του κειμένου. Θα πρέπει να εργαστούμε λοιπόν σκληρά επ' αυτού. Τώρα για την εκδήλωση της ΟΚΕ. Θα συζητήσουμε περισσότερο αύριο για τη σύμβαση και χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι η γνωμοδότηση επιθετής θα αναφέρεται συγκεκριμένα στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ως έγγραφο αναφοράς για οποιαδήποτε ολοκληρωμένη προσέγγιση στο ζήτημα της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. και άρθρο 12. Αν πάμε στο άρθρο 12, έχω ενώπιόν μου το κείμενο, αναφέρεται εκεί στις υποχρεώσεις. Περισσότερο έχουμε το άρθρο 3 που ορίζει το φύλλο, ενώ στο άρθρο 12 αναφέρονται και τα στερεότυπα στην παροχή προστασίας ε, στις πιο ευάλωτες γυναίκες, στους πιο ευάλωτες πληθυσμούς, εκεί αναφέρονται οι γυναίκες, ε, διάφορες ομάδες ε, όπως οι ομοφιλόφιλοι, ενθυλικοί κτλ. Ξέρετε, δεν αφήνουμε τους ανθρώπους να πεθάνουν επειδή μπορεί να είναι ομοφιλόφιλοι φιλική λοιπόν ο ορισμός του φίλου είναι μία από τις καινοτομίες της σύμβασης και μπορεί να θέτει πρόβλημα για ορισμένα κράτη-μέλη. Ήταν ε, αυτό το επίκεντρο της συζήτησης στην Πολωνία. Ξέρετε, δεν ε, μπορεί να υπάρξει επιφύλαξη για το άρθρο αυτό. Βέβαια, μπορεί να θέτει πρόβλημα σε ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά ελπίζω ότι θα το ξεπεράσουν ε, και θα δουν τι υπάρχει πίσω από τον ορισμό του φίλου και πίσω από το άρθρο αυτό και θα καταλάβουν ότι εδώ μιλάμε για την προστασία και την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που μπορεί να είναι ακόμη πιο εκτεθειμένοι στη βία επειδή είναι ακριβώς αυτοί που είναι. Και η παροχή προστασίας ε, στους ανθρώπους αυτούς ε, δεν πρέπει να εξαρτάται για το αν είναι από το αν είναι μετανάστες, αν είναι ομοφιλόφιλοι, αν είναι έγκυες γυναίκες. Έτσι λοιπόν εδώ μιλάμε περισσότερο για ανθρώπινα δικαιώματα παρά για την προστασία του τάδε ή το δίνα ε, για το αν είναι λεσβία, μια συγκεκριμένη κάνει είναι έγκυος, κάποια μετανάστρια κτλ. Ας το δούμε από τη σκοπιά του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ότι κάποιος πρέπει να προστατεύεται από τη βία επειδή είναι δικαιωμά του. Επίσης, για τα καταφύγια, αναφέρθηκε ανάγκη να έχουμε περισσότερα. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Είναι μακροσκελής η σύνδεση, έχουμε πολλά άρθρα. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη, η οποία αναφέρεται στα καταφύγια Πρέπει να υπάρχουν καταφύγια και πρέπει να υπάρχουν και τηλεφωνικές γραμμές 24 ώρες, 24 ώρο, όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στις αγροτικές περιοχές. Και θέλω να σας αναφέρω ένα σημαντικό μήνυμα. Είναι πλήρες το κείμενο. Ευχαρίστω να σας δώσουμε βοήθεια επί συγκεκριμένων άρθρων και διατάξεων αν το χρειάζεστε. Όμως το πιο σημαντικό είναι τώρα να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το κείμενο και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητε κυρώσει για την εφαρμογή του. Γιατί όπως σας είπα παραμείνει ένα ωραίο νομικό κείμενο δεν θα ωφελήσει καθόλου τις γυναίκες που είναι θύματα βίας εκεί έξω. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει λοιπόν από τη δική μας πλευρά, αναφέρεται και μία παρέμβαση στην Ουγγαρία, θα ήταν καλό, θα ήταν καλό να απαντήσουμε σε αιτήματα των κρατών μελών από τον περασμένο Οκτώβριο. Όταν εγώ έλαβα αυτό το τμήμα έχουμε οργανώσει πάνω από 100 εκδηλώσει. Οργανώθηκαν είτε από εμά είτε από άλλους θεσμού από Εθνικά Κοινοβούλια ή αρχές. Και είμαστε μόνο δύο άτομα που δουλεύουμε επί της σύμβασης αυτής. Όμως ε, θα κάνουμε τα δυνατά μας. Ε, έχουμε ένα πολύ καλό δίκτυο εμπειρογνωμόνων ε, που θα προσπαθήσει να στείλει πληροφορίες στα κράτη-μέλη για να εξηγήσουμε τη φιλοσοφία των άρθρων της σύμβασης στα κράτη-μέλη. Και φυσικά βασιζόμαστε και στη δική σας βοήθεια για να προωθήσουμε τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα λέγοντας ότι είμαστε ευγνώμονες για την όλη συζήτηση, για όλα τα σχόλια που ακούστηκαν. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο να διαπιστώνει κανείς πόσο αφιερωμένα και αφοσιωμένα είναι τα, τα μέλη ε, σε κάποια θέματα όπως αυτό. Αισθάνομαι περήφανος ως πρόεδρος και πάντοτε όταν έχουμε κάποιο προσκεκλημένο, πάντοτε λέω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεσμεύεται σε στενή συνεργασία μαζί σας για αυτό το σκοπό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί εδώ αυτή η συνεργασία έχει γίνει ήδη πράξη. Βεβαίως υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν ακόμη και βεβαίως θα προχωρήσουμε και σε αυτά. Να μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται από την ε, άνηση, από τον άνηση συσχετισμό δυνάμεων που πάντοτε υπάρχουν και πάντοτε κάποιοι έχουν μεγαλύτερη εξουσία την οποία ασκούν σε κάποιους άλλους. Υπάρχει λοιπόν ανισότητα ε, στην κοινωνία μας και υπάρχει ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και πολύ ορθά είπε η κυρία Στρέλα ότι η καλή βάση θα ήταν Πρώτα απ' όλα να υπάρχει μια τέτοια οικονομική άνεση ώστε να μπορούν οι γυναίκες να είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Από εκεί μπορεί να ξεκινήσει κάτι καλά. Όταν μιλάμε για συσχετισμό δυνάμων και εξουσιών, όπως είπε η κυρία Τόμσον, επαναρχόμαστε στο ζήτημα κατά πόσον είναι άρρωστος ε, ψυχικά ένας άνθρωπος που χτυπάει τη γυναίκα του. Αλλά λέει ε, ο αντίλογος, μα δεν πάει να χτυπάει όλο τον κόσμο, δεν χτυπάει τον ε, ταξιτζή ή τον οδηγό του λεωφορείου ή οποιοδήποτε άλλο. Χτυπάει τη γυναίκα του. Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν για την παρουσία σας στην ε, σημερινή μας συζήτηση. Ε, φαίνεται και ότι στην πολύ καλή σχέση που έχετε με την Επιτροπή μας και φαίνεται και από το εγχειρίδιο που μας δώσατε ε, ώστε να μπορέσουν ε, μέσω αυτού του φυλαδίου και οι συνάδελφοι να περάσουν πιο πέρα το μήνυμά σας και εμείς ως ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να περάσουμε αυτό το μήνυμα στην κοινωνία. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δουλέψουμε και σε πολλά άλλα μέτωπα. Κυρίως να ασκήσουμε πίεση στις χώρες μας να κυρώσουν τη σύμβαση. Δύο μέτωπα, αν θέλετε, δύο μάχες που μπορούμε να δώσουμε παράλληλα. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε να κυρώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτή τη σύμβαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Vi eh, Ας συνεχίσουμε με τα σημεία της σημερινής διάταξης. Ουσιαστικά μας μένει το τελευταίο για τη σημερινή μας συνεδρία, στο σημείο 16. Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2011.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 διότι υπάρχει μια έκτη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας, οπότε μου ζήτησε να διαβάσω ένα σημείωμά τη για αυτή την ε, γνωμοδότηση που συνέταξε σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο του 2011 και σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Θα σας, προετοι... θα σας παρουσιάσω ένα σχεδίο γνωμοδότηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο 2011 και την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική για μα, γιατί κάθε χρόνο μα παρουσιάζει νέα δεδομένα σε σχέση με την πρόοδο που έχει σημειωθεί με την παναχώρηση στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών και αξιών όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η ισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών μεταξύ άλλων. Σε αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, ήθελα να παρουσιάσω κυρίως ε, τέσσερις ε, θεματικές που είναι ζωτική σημασίας για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται καλύτερα υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών. Γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα μιλάμε επίσης και για τα δικαιώματα των γυναικών. Καταρχήν ήθελα να επιμείνω στην σημασία της συστηματικής ε, συμπερίληψης της ισότητας ε, των δύο φύλων και της πρόθεσης των δικαιωμάτων των γυναικών ε, στο διάλογο που έχει η Ένωση με τις τρίτες χώρες, κυρίως στα πλαίσια συμφωνιών, οικονομικών συμφωνιών ή συμφωνιών σύμπραξης. Επίσης, ε, είναι σημαντικό ο σου εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συμπεριλάβει στις προτεραιότητες της θητείας του την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την πρόθεση της αυτονόμησής τους. Τρίτον, είναι σημαντικό να επιμείνουμε στην αναγκαιότητα να συμπεριλάβουμε μια προσέγγιση ε, για την ισότητα των δύο φύλων σε όλα τα στρατηγικά έγγραφα, τα σχέδια δράσης και σε κάθε άλλο εγγραφό ε, εξωτερικής δράσης της Ένωσης προκειμένου να εγγυθούμε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την πλήρη συμμετοχή του στην κοινωνία. Τέλος. Είναι επίσης απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα των Δύο Φύλων να ενισχυθεί και στο μέτρο του δυνατού να παρέχει περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα προκειμένου και τα υπόλοιπα νομοκτήματα και τα μέσα εξωτερικής δράσης να είναι όλα και πιο αποτελεσματικά. Αν υπομονώ, η συνάδελφός μου η Μαρία δηλαδή, να ακούσω ε, όλα τα σχολιά σας, θα περιμένω μάλλον τα σχολιά σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις προτάσεις σας. Σας ευχαριστώ. Ehm. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ε, έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Α, παρακαλώ, κυρία Μαρβάη έχει το λόγο. Ναι, Ως ε, πρώην μέλος της αρμόδιας Επιτροπής των Μένων Εθνών για αυτό το ζήτημα, ξέρετε, ε, έχω μια κάποια ανησυχία. Πώς άνδρες και γυναίκες μπορούν να γνωρίζουν ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την επιτροπή, όπως εκπροσωπούνται, ποια... ποιες είναι οι ανάγκες και επιθυμίες των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται να ακούσουμε τη φωνή, πιστεύω, των ανθρώπων. Να ακούσουμε αυθεντικά τις φωνές των γυναικών, τις ακάστοτε κοινωνίας ή χώρας που μας απασχολεί. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, λέει ομιλήτρια, ε, να μην γίνονται συζητήσεις παράλληλα την ώρα που συνεδριάζαμε, ε, διότι ε, σταματούν τη σκέψη μας. Αν μπορούν, όσοι έχουν συζητήσει, να τις κάνουν εκτός αιθούσες. Λοιπόν, να έχουμε επαφέ με τις ίδιες τις γυναίκες με τις μη κυβερνικές οργανώσεις για να μπορέσουμε να είμαστε πιο σίγουροι ότι έχουμε κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των γυναικών στην εκάστοτε κοινωνία. Παράδειγμα, μουσουλμάνες. Εμείς εδώ, σε μια δυτική κοινωνία, ίσως πιστεύουμε ότι στο μουσουλμανικό κόσμο η γυναίκα είναι υποταγμένη. Πράγματα και πρακτικές, κατά τη γνώμη μας, είναι κακά, αρνητικά. Αντίθετα όμως υπάρχουν ισχυρά φεμινιστικά κινήματα σε μουσουλμανικές χώρες και πολλές φορές οι γυναίκες στις χώρες αυτές πιστεύουν τα πράγματα διαφορετικά. Είναι σημαντικό να έχουμε μια α, πλειάδα απόψεων και όσο πιο πολλές απόψεις έχουμε, τόσο πιο καλή εικόνα της πραγματικότητας θα μπορούμε να αποκομίσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια αυτοπεποίθηση ότι εμείς μόνο κατέχουμε την αλήθεια, ότι γνωρίζουμε ακριβώς τις ανάγκες των γυναικών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω τώρα μπορώ να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν δίνετε το λόγο. Οπότε, η κυρία Μπάστος, μήπως θέλει να κάνει ένα τελικό σχόλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τη συνάδελφο και την τοποθέτησή της, την οποία θα διαβιβάσω και στην εισηγήτρια, καταγράφοντας ανησυχίες που ακούστηκαν στην αίθουσα. δεν έχουμε την παρουσία εκπροσώπου της Ευρωπαϊκή Επιτροπής σήμερα, αλλά πιστεύω ότι σε μεταγενέστερη συζήτηση για την ίδια έκθεση θα έχουμε παρουσία της Κομισιόν. Κατά τα λοιπά θα διαβιβάσω τα υπόλοιπα στη Μαρία Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ. Yes, please, you have the floor. Έχετε το λόγο. Ε, δεν είμαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένα θέματα τα οποία έχουν ε, συζητηθεί. Καταρχήν, Συμφωνώ απολύτως με την ε, αρχική ε, δήλωση της κυρίας Μπάστος ότι οι γυναίκες ανοίγουν το δρόμο του ανθρωπίνου γένους και ε, αντιλαμβάνομαι πλήρως την άποψη της κυρίας Γκαμπριέλ θα περάσω το μήνυμά σας στον κύριο Σταύρο Λαμπρινίδη όπως και τα σχόλιά σας και την αίτηση να φροντίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όντως ενδιαφέρεται ούτως ή άλλως πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Είχαμε μία συνάντηση στη, της Διευθύνσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον κύριο Λαμπρινίδη και το θέμα που έθιξε ε, ήταν ε, ότι ένα από τα θέματα στα οποία επικεντρώνεται ε, ήταν ένας γύρος του τραπεζού για να ρωτήσει τι μπορεί να γίνει σε γενικό επίπεδο για βελτίωση της κατάστασης των γυναικών Οπότε ε, προφανώς θα περιλάβει τα δικαιώματα των γυναικών στο στρατηγικό μας έγγραφο και ξέρω ότι η απόφαση του Συμβουλίου τον Ιούνιο εφέτος αναφέρεται συγκεκριμένα στα δικαιώματα των γυναικών που αποτελούν ένα βασικό ε, στρατηγικό ενδιαφέρον ε, της ευρωπαικης ενωσης Ενώσεως. Υπάρχουν ε, τέσσερις-πέντε τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και ιδιαιτέρως η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη μπορούν να κινηθούν για να βελτιώσουν ε, και να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και τέλος ο, ε, η ύπατος επιτετραμένη ε, θίγει το θέμα αυτό και με τους εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών σε άλλες χώρες και με τις γυναίκες συγκεκριμένως ιδίω όταν υπάρχουν διάλογοι και διαβουλεύσεις με τρεις χώρες και έχω ε, συμμετάσχει κατά την τελευταία πενταετία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ένα θέμα που προκύπτει τακτικότατα στους διαλόγους και στις διαβουλεύσεις μας. Τέλος, όσον αφορά τις ε, γυναίκες με την διαχείριση της κρίσεως, θεωρούμε ότι είναι ένας από τους πυρήνες δράσεώς μας. Ακούμε τις ομάδες γυναικών για την πρακτική αξία και μπορώ έτσι να αναφερθώ εις την εργασία μου διότι οι γυναίκες μπορούσαν να μας πούν που φυλασσόντουσαν τα όπλα και κατά αυτόν τον τρόπο να αυξήσουν την τη δραστηριότητά μας οπότε βλέπετε ότι ε, αν ε, όντως περιλαμβάνουμε ε, τις γυναίκες υπάρχει μεγάλο όφελος η κυρία Γκουρμάη με συγχωρείτε ήρθα καθυστερημένη αλλά ιδίως από όταν άκουσα τα σχόλιά σας είναι πολύ βασικό που είσαστε και εσείς γυναίκα και καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε όταν συζητάμε το θέμα αυτό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι κάθε άστον ε, έχει θεωρήσει πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και ότι έχουμε όλο και περισσότερες γυναίκες στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Δεν επαρκούν μεν, αλλά προχωράμε. Είναι βασικό θέμα. Ευχαριστώ τον εισηγητή και αυτό που είναι βασικό είναι ότι έχει λάβει υπόψη όλα τα βασικά θέματα. Είναι βέβαια σημαντικό ότι συμπεριελήφθη τον χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το θέμα των γυναικών κατά τρόπον ώστε να υπάρχει ισότητα αντιμετώπισης σε όλες τις εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά τον κύριο Σταύρο Ναμπρινίδη, ο πρώην ε, Έλληνας Ευρωβουλευτής και συνάδελφος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι πολύ προοδευτικό στον τομέα αυτό, έχει αναλάβει αυτό το σημαντικό ε, ρόλο, ιδίως όσον αφορά το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει επιπλέον η συγκήτρια να λάβει υπόψη την Αραβική Άνοιξη όπου οι γυναίκες ήταν ε, στις πρώτες γραμμές της ε, ε, επαναστάσεως το ίδιο και στην Ουγγαρία στη δεκαετία του 90 οι γυναίκες είχαν προηγηθεί και στη συνέχεια δεν είδαμε να καλύπτουν τόσες πολλές θέσεις παρόλο που σε ορισμένα κράτη έχει βελτιωθεί η ποσόστοση για εκπροσώπηση των γυναικών. Ε, πρέπει λοιπόν να τονίσουμε τον ρόλο των γυναικών και την συμμετοχή τους ιδίως ε, όσον αφορά τη διαδικασία λήψεως αποφάσεως, αλλά υπάρχει κρίση και οι γυναίκες έχουν ε, ένα ειδικό ρόλο. Δεν σημαίνει ότι οι άντρες τη διαχειρίζονται καλύτερα, αλλά βλέπετε ότι στην κρίση έχουν συμμετάσχει πολύ περισσότερες γυναίκες για να λύσουν ε, το θέμα της κρίσεως. Αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες οι γυναίκες αυτές, ας τους αφήσουμε να κάνουν τις ε, ε, δουλειά τους και ουσιαστικά πιστεύω ότι στα κοινά μας θέματα θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία για τα θέματα των γυναικών. Ευχαριστώ. Αυτό ολοκληρώνει τη συζήτηση. Και τώρα μπορώ να σας πω ότι θα πρέπει η ε, τροπολογίες να έχουν υποβληθεί μέχρι τις, ε, ε, ε, τις 29 Ενάτου στις 5 το απόγευμα στην Επιτροπή θα ψηφίσουμε 18 στην Ολομέλεια 10 11 και ε, τώρα μπορούμε να πάμε στο τελευταίο θέμα της ημερησίας διατάξεως, το, την προσεχή συνεδρίαση που θα είναι 10 Οκτωβρίου, 9 με 12.30 και 3 με 6.30. Ε, αυτό ολοκληρώνει τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ όλους και ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα.